Ξαναξεκινάμε λοιπόν την σύνοδο μας ε, πληροφοριακά να σας πω ότι ο κύριος Δημήτρ Στογιάνοφ μου ζήτησε ε, να επικαλεστεί την κοινοβουλευτική του ασυλία ε, με την ευκαιρία μιας